Βλέπω ότι η κυρία Κρέιτον δεν έχει έρθει ακόμα και γι' αυτό θα έλεγα να ξεκινήσουμε με τον κύριο Μπαρόζο. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, τακτικά επισύρω την προσοχή σας στην έλλειψη πολιτικών σχέσεων του Κοινοβουλίου με τον ε, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ε, γράψα να, για να προσκληθεί σε αυτήν την προκαταρτική συνεδρίαση, ούτω ώστε να, ε, καθώς συζητούμε τις ε, νομοθετικές πτυχές με το ε, Συμβούλιο και τις οικονομικές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με την εφαρμογή του άρθρου 15 της συνθήκης και λυπούμε ότι η προσπάθεια που κάναμε με τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας εχθές έπρεπε να το κάνουμε και με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Λυπούμε που δεν να έγινε αποδεκτή η πρόσκλησή μας. Ε, την παραμονή μάλιστα ενό Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πολύ σημαντικού όπου θα διαπραγματευτεί το Συμβούλιο τις δημοσιονομικές ε, προοπτικές. Πρέπει να υπάρξει πολιτική σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ελπίζω κύριε Πρόεδρε κάποια μέρα και εσείς ε, θα συμμετέχετε σε όλες τις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα παρίσταται στις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, κύριε Ρουντή, φαντάζομαι μιλάτε για τον κύριο Φαν Ρομπέι ο κύριος Φαν Χομπέι είναι μόνιμος προσκεκλημένος ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά ο ίδιος ε, πιστεύει ότι οι συνομιλητές του είναι οι κυβερνήσεις και όχι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Του έχω πει επανειλημμένα ότι εμείς ε, έχουμε διαφορετική άποψη αλλά ε, γνωρίζω στην πολιτική σας ομάδα ε, αρκετούς ευρωβουλευτές ε, που βρίσκονται πολύ κοντά στον κύριο Βαν Χομπέου. Ίσως λοιπόν μπορείτε να ασκήσετε εσείς πίεση και να του πείτε μάλλα επιτέλους στο Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι αυτό νομίζουμε ότι αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο. Εγώ το το λέω συνέχεια. Αλλά βέβαια πρέπει να σας πω επίσης ότι σε καθαρά τυπικό και νομικό επίπεδο ο συνομιλητής του Κοινοβουλίου δεν είναι ο κ. Βαν Χομπέου αλλά ο προεδρεύων του Συμβουλίου. Ε, παρόλα αυτά αυτά οι ε, αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων πιστεύουν ότι ο συνομιλητή του είναι ο κ. Βαν Χομπέ. Βλέπετε λοιπόν ότι όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ακόμα πρέπει να διευκρινιστούν πολλά πράγματα. Ε, ο κ. Σφάμποντα, κοιτάξτε, στηρίζω προφανώς ανεπιφύλακτα αυτό που ελέγχθη, αλλά μήπω αυτά που είπατε σημαίνουν ότι οι διαπραγματεύσει ε, που θα διεξαχθούν για τον προπολογισμό θα πρέπει να γίνουν με την Ιρλανδική Προεδρία. Γιατί αν ο συνομιλητή μα δεν ο κ. Βαν Χομπέ, τότε προφανώ συνάγω ότι η συνομιλητής μα είναι Ιρλανδική Προεδρία. Πρόεδρο κύριε Σφόποντα, η συνθήκη είναι σαφής. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αύριο και την Παρασκευή θα αποφασίσει για τη διαμόρφωση της πολιτικής βούληση, Δηλαδή ε, το ε, καθαρά τυπικό πλαίσιο με βάση το άρθρο 312 ε, του, της συνθήκης ο, ο προεδρεύων. Ε, βλέπετε μόλις τώρα μπαίνει στην αίθουσα. Εγώ να σας πω ότι ο συνομιλητής μας στις διαπραγματεύσεις είναι ο Πρωθυπουργό κύριος Κέννη. Κύριε Σβόμποντα, νομίζω το γνωρίζετε αυτό, το έχω πει εξάλλου επανειλημμένα στη διάσκεψη των Πρόεδρων. Και παρεπιπτόντος ε, το έχω αναφέρει και στην τετραμερή συνάντηση ότι ο συνομιλητής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κανονικά είναι Ιρλανδική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με συγχωρείτε, είναι Ιρλανδική Προεδρία. Τις διαπραγματεύσει όμως τις διεξάγει ο κύριος Βαν Χομπέι. Ε, στο σημείο αυτό η συνθήκη είναι ασαφής και νομίζω ότι πρέπει να ε, διευκρινιστεί το θέμα. Αυτά. Ε, κατά τα άλλα, κύριε Κρέιτον, χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθατε και θα μου επιτρέψετε να σας δώσω το λόγο για τη δήλωση του Συμβουλίου σχετικά με την προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη.